Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie wiceprzewodniczącego. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στη δήλωση τη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι εξωτερικέ υποθέσει και την ασφάλεια για την κατάσταση στη Λευκορωσία. Θα ήθελα να τη δώσω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε τα γεγονότα μετά από τις εκλογές της Λευκορωσίας 19 ε, Δεκεμβρίου μα σώκαραν όλους. Η βία των αρχών κατά των πολιτών οδήγησαν σε ανησυχία και καταδίκη από όλο τον κόσμο και υποφαινόμενοι και οι συνάδελφοί μας συνάντησαν με πολλούς από εκείνους που επλήγησαν μεταξύ της αντιπολίπωσης της κοινωνίας των ε, πολιτών, των εκπροσώπων των φυλακισμένων και γενικά της κοινωνίας για να εκφράσουμε την συμπάθειά μας, την αλληλεγγύη μας και να τους ακούσουμε. Τώρα όμως έχει έρθει πια η στιγμή για να δράσουμε. Ε, κτιμώ το γεγονός ότι μέλη ε, του Σώματος μπορούν να συμβάλλουν στη σκέψη για το θέμα αυτό. Και ο συνάδελφος ε, Επίτροπος ε, Φούλερ μπόρεσε να παρουσιάσει τις πρόσφατες ε, σκέψεις μας στην Επιτροπή ΑΦΕ την περασμένη εβδομάδα. Ε, περιμένω με ανησυχία την, ε, το ψήφισμά σα ε, που προέρχεται από τη δική σα εργασία. Ε, πρέπει οπωσδήποτε να δράσουμε. Το θέμα είναι πήγον. Ε, ασχολήθηκα με μέλη τους, της αντιπολίτευσης, με ε, συγγενείς των κρατουμένων και τον ε, Πρωθυπουργό Ματίνοφ. Αυτά που έδειξαν ότι πρόκειται για μια προσβολή του δικού μας οράματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις βασικές αρχές και τη δημοκρατία. Η εκλογική διαδικασία γενικά υποσκάφθη από την κράτηση εκπροσώπων της κοινωνίας των πρατων και της αντιπολίτευσης. Οι αξιολογήσεις και της ΟΑΣΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σύμφωνες. Πολλοί από αυτούς που κρατήθηκαν έχουν απελευθερωθεί. Παρ' αυτά, μια μεγάλη ομάδα, 30 άτομα, αντιμετωπίζουν ακόμα την, ε, την δυνατότητα ε, κράτησης για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μεταξύ αυτών ήταν και ορισμένοι υποψήφοι για την Προεδρία. Έχω κάνει έκκληση για την άμεση απελευθέρωση όλων εκείνων που κρατούνται για πολιτικούς ε, λόγους καθώς επίσης και το να ξανανοίξει το γραφείο σα στην ε, ΟΑΣΕ συγγνώμη στο Μίνσκ στην συνάντησή μου με τον ε, Υπουργό Εξωτερικών Μαρτινόφ τόνισα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένει άμεση απάντηση από τις αρχές της Λευκορωσίας στα αιτήματα της διεθνούς κοινότητας. Καθορίζοντα τα επόμενα μα βήματα, θα πρέπει να βασιστούμε σε βασικέ αρχέ. Η πρώτη από τι αρχέ αυτέ είναι ότι η ασφάλεια ε, ε, και η, και η, και η για τους ε, αντιφροντούντες θα πρέπει να είναι η πρώτη μας μέρημνα. Δεν μπορούμε να απομονώσουμε τους πολίτες. Επίσης θα πρέπει να σεβαστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες που είναι ένα βασικό τμήμα τις εταιρικέ σχέσεις που έχουμε και τις κοινέ αξίες που συμμεριζόμαστε με τους ε, πλουσίων μας εμάς εταίρους. Θα συνεργαστούμε με τους εταίρους αυτούς όπως το κάναμε και με τη ΣΥΠΑ για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις εξελίξεις στην Λευκορωσία. Αυτό σημαίνει εν καταλήξει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλους του διάβλους για να δράσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά με ένα σωστό μήνυμα έναντι των αρχών της Λευκορωσίας χωρίς να απονομήσουμε τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών. Η αντίδρασή μας θα πρέπει να είναι ισορροπημένη. Αφενός θα πρέπει να δούμε τη δυνατότητα εστίασης μέτρων προς τις αρχές ε, της Λευκορωσίας. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να έχουμε έντονο διάλογο με και υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε την υποστήριξή μας των μη κυβερνικών των το των ΜΜΕ των φοιτητών και να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας για να αυξήσουμε την κινητικότητα των πολιτών που θέλουν να στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βράχει πρόθεσμα θα πρέπει να επαναφέρουμε την απαγόρευση ε, ταξιδίου για τον ε, Πρωθυπουργό Λουκασιανκό και να διευκρίνουμε μάλιστα αυτή τη δράση. Θα αυξήσουμε έτσι αυτή τη δράση σε συνεργασία με την Κομισιόν για να προωθήσουμε μέτρα υπέρ των ΜΜΕ, των μη κυβερνικών των οργανώσεων και των φοιτητών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατά νου να δώσει υποτροφίε για φοιτητέ που έχουν εκδοχθεί από τα πανεπιστήμια και ελπίζω να μπορέσουμε να προωθήσουμε τη δυνατότητα αυτή και να υπάρχουν και επαρκεί πηγέ και από αλλού, δηλαδή και από τα κράτη-μέλη. Αναφέρθηκα ήδη στο θέμα της κινητικότητας και έχω εδώ κατά νου κυρίως τις διευκολύνσεις για τη θεωρήση Θα θέλω να ενθαρρύνω τα ε, προξενία των κρατών μελών στο ΜΙΣΚ να διευκολύσουν την χορήγηση θεωρήσεων προς όφελος των, των πολιτών. Αυτά είναι βέβαια ε, ορισμένα μέτρα που θα πρέπει να εξεταστούν στις 31 Γενωρίου από το Συμβούλιο Εκτορικών Υποθέσεων. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε, θα πρέπει να επανεξετάσουμε ορισμένες πτυχές των σχέσεών μας με την Λευκορωσία. Θα πρέπει να συνεργαστούμε και με τους άλλους διεθνείς ε, εταίρους μας για την Λευκορωσία και με την ίδια τη Λευκορωσία και να συνεργαστούμε με τους ε, εταίρους μας της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Επίσης όσον αφορά την συνεδρίαση των προστασιών μας στη κοινωνία πολιτών και στους πολιτές. Τέλος, είχαμε ξεκινήσει πέρσι ένα σχέδιο για την ε, καταγραφή των σχέσεών μας τα επόμενα χρόνια. Δεν έχουμε καταλήψει αυτό το προσωρινό ε, κοινό πρόγραμμα, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα ξανατοποθετηθεί μετά τα γεγονότα. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο εργαζόμαστε και θα ακούσουμε με ενδιαφέρον τι απόψει των μελών του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε. Και τώρα εκ μέρου των πολιτικών ομάδων θα λάβουν το λόγο διάφοροι ομιλητέ. Ο κύριο Προτάσοβιτ πρώτα για το ΕΛΚ. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λίδη Άστον. Πρέπει να σας πω ότι οι διεθνείς παρατηρητές δεν είχαν καμία αμφιβολία και δεν πρέπει να αποκτήσουμε εμείς αμφιβολίες. Οι τελευταίες εκλογές δεν ήταν δίκαιες ούτε τιμίες. Δεν ήταν λοιπόν δίκαιες και σαν αποτέλεσμα αυτού είναι ότι η πολιτική που εφαρμόσαμε σε σχέση με τις αρχές της Λευκορωσίας η πολιτική μας πρέπει να διακοπεί, πρέπει να αλλάξουμε προσέγγιση. Δεν είναι ώρα τώρα να κάνουμε τα ίδια πράγματα όπως συνήθως ήρθε η ώρα για νέες αποφάσεις, νέα πολιτική αποφασιστικότητα σε σχέση με το καθεστώς του Λουκασάνικο και για κυρώσεις είναι όριμη η ώρα. Ε, πολιτικές κυρώσεις τη Βίζα, αλλά δεν πρέπει να αποκλείσουμε και τις οικονομικές κυρώσεις. Δεν πρέπει βέβαια να υποβαθμίσουμε τη ζωή του λαού, αλλά θα πρέπει να τολμήσουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις. Ακόμη θα πρέπει να σκεφτούμε να ανακαλέσουμε τη σχέση της Λευκορωσίας με τη δυτική πλευρά. Οι νικητές των εκλογών ουσιαστικά είναι η δημοκρατική αντιπολίτευση της Λευκορωσίας. Πρέπει συνεπώς να υποστηρίξουμε αυτή την αντιπολίτευση και να αποκτήσει κάποια εκπροσώπηση εδώ ή στις Βρυξέλλες. Αυτή η εκπροσώπηση της αντιπολιτευσής θα μπορούσε να είναι η εκπροσώπηση της χώρας στον κόσμο ολόκληρο. Θα επίσης κάνω έκκληση να ε, αποφυλακιστούν όλοι οι διαδηλωτές, οι δημοσιογράφοι, οι υποψήφοι, όλοι πρέπει να αποφυλακιστούν πριν ακόμη σκεφτούμε να ξαναρχίσουμε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Ο κύριος Μπεγκίνεν εκ μέρους των σοσιαλιστών τώρα. Και θα ήθελα εδώ να πω σε σχέση με τις εκλογές στην Λευκορωσία και τις χαμένες ευκαιρίες την δυνατότητα να ακολουθηθεί η δημοκρατική πορεία. Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια πολιτική του συμβιβασμού βήμα προς βήμα ή της προσαρμογής βήμα προς βήμα. Υπάρχουν κάποια τέτοια στοιχεία. Αν θέλουμε όμως ε, να ανατρέψουμε αυτήν την πολιτική πρέπει να είμαστε προσεκτικοί διότι η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, οδήγησε στο ότι η Λευκορωσία μέσα στο πλαίσιο των προεδρικών εκλογών κατάφερε να σημειώσει κάποιες προόδους. Ένα, μια ένδειξη αυτών των, αυτής πρόοδου ήταν ότι κατά τη νύχτα των εκλογών πολύ περισσότεροι πολίτες κατέληξαν σε, στους ε, με διάφορες εκδηλώσεις από ό,τι αναμενόταν. Με άλλα λόγια ήταν μεγαλύτερη η ελευθερία που μπορούσε κανείς να παρατηρήσει όσον αφορά τους πολίτες αυτούς. Εφ' θα πρέπει να είμαστε αρκετά σαφείς και στεναροί, αποφασιστικοί. Έχω υπόψη εδώ το αίτημα απέναντι στη Λευκορωσία να απελευθερωθούν όλοι οι κρατούμενοι. Και η δίωξη όλων των διοκόμενων και κρατούμενων να σταματήσει αμέσως των ατόμων εκείνων που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις ή που είχαν εμπλοκή στις διαδηλώσεις αυτές. Πρέπει να είμαστε εδώ πάρα πολύ σκληροί και να μην δείξουμε κανένα συμβιβασμό και να μην υπαναχωρήσουμε διατυπώνοντας με σαφήνεια τα αιτήματά μας. Τι μπορούμε όμως μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να κάνουμε. Αφενός πρέπει να αποφύγουμε να απομονωθεί η Λευκορωσία εκ νέου. Οι εκπρόσωποι εκεί της κοινωνίας των πολιτών έχουν σαφώς τονίσει και έχουν αναφέρει ότι μια απομόνωση της Λευκορωσίας θα είναι απομόνωση των πολιτών ταυτόχρονα. Και αυτό πρέπει να αποφευθεί. Όσον αφορά την πολιτική μας έναντι της Λευκορωσίας, θα πρέπει αυτή να αλλάξει και είναι αναγκαίο να αλλάξει. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες της Λευκορωσίας θα αποκομίσουν τα μέγιστα ωφέλη και όχι μόνο οι πολίτες αλλά επίσης και τα μέσα της ενημέρωσης και το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών. Αν αλλάζαμε λοιπόν τις πολιτικές μας, την πολιτική μας τότε θα ήταν εφικτό να διεξαχθούν και δημοκρατικές εκλογές. Θα πρέπει με άλλες τρίτες χώρες να συνεργαστούμε και με την Ρωσία και την Ουκρανία προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει ως Ευρωκοινοβούλιο να δραχθούμε των ευκαιριών της ανατολικής γειτονικής σχέσης, της σχέσης γειτνίασης, ώστε αυτή η εταιρική σχέση να συνεισφέρει για τον εκδημοκρατισμό εκεί. Ευχαριστώ. Έχουμε μια μπλε κάρτα, κύριε. Είστε έτοιμος να απαντήσετε. Ο κύριος Μιγκάλσκι. Συνάδελφε, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, έχω μόνο 30 δευτερόλεπτα. Ίσως υπήρξε κάποια παρεξήγηση. Εγώ κατάλαβα ότι σύμφωνα με εσά οι διαδηλώσει αυτές μετά τις εκλογές, αυτή η διαδήλωση δηλαδή, που ήθελα να διαμαρτυρηθεί κατά των διαφόρων παραβιάσεων που έγιναν στις εκλογές, κατά της εκλογικής νοθείας, θεωρούνται σαν το κίνητρο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή της κατάστασης. Θέλω να ξέρω, αυτό είπατε, γιατί αν είπατε κάτι τέτοιο δεν μπορώ να δεχτώ αυτή την τοποθέτηση. θα πρέπει να πω ότι ήταν αρκετά σαφής η τοποθέτηση και καμιά φορά στη διαρμηνία οι λεπτότητες ε, είναι ε, κάτι, ένα στοιχείο το οποίο χάνεται ε, και έχει αλλάξει η κατάσταση στη Λευκορωσία μια και όλο και περισσότεροι πολίτες αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της δημοκρατίας βλέπουν οι πολίτες την ανάγκη να αγωνιστούν για τη δημοκρατία στις εκλογές υπήρχαν πολύ περισσότεροι πολίτες στους δρόμους της πόλης του Μίνσκ, πολύ περισσότεροι από ό,τι αναμενόταν. Και αυτό όχι μόνο σε σχέση με το πολιτικό καθεστώς. Ευχαριστώ. Πιθανότατα κάτι δεν πέρασε. Υπάρχει πρόβλημα τεχνικό με την ε, αγγλική μετάφραση. Παρακαλώ, γίνει ένας έλεγχος. Δεν ακούγονται τα αγγλικά. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Δεν περνάει η διερμηνία bench. Κοιτάξτε, παρεξήγηση υπήρξε. Προσπαθώ πάντα να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Ίσως, άμα είναι ευαίσθητο το θέμα, θα πρέπει να εκφράζομαι σε άλλη γλώσσα. Τι προσπαθούσα να διαβιβάσω. Βελτιώνεται η κατάσταση. Γιατί το λέω όλο και περισσότεροι στη Λευκορωσία καταλαβαίνουν ότι η Λευκορωσία χρειάζεται τη δημοκρατία και όλο και περισσότεροι καταλαβαίνουν ότι πρέπει να πολεμήσουν για την δημοκρατία στη Λευκορωσία. Γι' αυτό είπα ότι θεωρώ σαν θετικό μήνυμα το γεγονό ότι τόσο πολλοί κόσμος πολύ περισσότερα από αυτά που περίμεναν οι οργανωτέ, ήταν στην ε, πλατεία, κατεβήκαν στην πλατεία. Ελπίζω τώρα να καταλάβατε τι θέλω να πω. Ευχαριστώ η κυρία Κριστίνα Όγιουλαντ για τους ελευθέρους δημοκράτες. Κύριε Πρόεδρε, κυρία είπατε εκπρόσωπο, ήταν καλό που ακούσαμε αυτά που είπατε. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτά που είπατε και είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να αντιδρά όσον αφορά τα προβλήματα στις ειδικές εκλογές στη Λευκορωσία. Μακάρι να είχαμε το θάρρος να είμαστε τόσο στεναροί και να ακολουθούμε τις αρχές μας και στην περίπτωση μιας γειτονική χώρας της Λευκορωσίας όπου η καταστολή της, της αντιπολίτευσης του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν γίνει κοινό τόπος. Η ε, επιδείνωση κατάστασης της δημοκρατίας στη Ρωσία ίσως να είναι ο λόγος για τον οποίο το Κρεμλίνο έχει αναγνωρίσει τις προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία και περιέγραψε τη βίαιη καταστολή σαν εσωτερικό θέμα υπόθεση της Λευκορωσίας. Τέτοια διαφορία όσον αφορά τη φρικτή κατάσταση στην Λευκορωσία είναι ένα σημαντικό μήνυμα των τάσεων στη Ρωσία. Κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ισχυρό ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει συγκεκριμένε κυρώσει οικονομικέ και για τι θεωρήσει διαβατηρίων που στρέφονται κατά του καθεστώτο του Λουκασέγκο. Είναι ζωτική σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί ενωμένη όσον αφορά αυτό το θέμα και τα κράτη-μέλη επίσης να σταματήσουν οι εσδήποτε διμερείς πρωτοβουλίες με τον Λουκασέγκο και το καθεστώ του. Θα πρέπει να αναστείλουμε την εταιρική σχέση, την ανατολική και άλλη συνεργασία μέχρι ό,τι οι πολιτικοί κρατούμενοι να απελευθερωθούν. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αυξήσουμε την υποστήριξη προς την κοινωνία των πολιτών τις μη κυβερνητικέ οργανώσει και τα ανεξάρτητα μέσα στη Λευκορωσία για να του προετοιμάσουμε για την ανοικοδόμηση της Λευκορωσίας μετά την κατάρρευση του Λουκασέγκο που ελπίζουμε ότι θα λάβει χώρα μέσω δημοκρατικών εκλογών. Γι' αυτό θα ήθελα να υποστηρίξετε ένα πανευρωπαϊκό φόρουμ για το μέλλον της Λευκορωσίας να διοργανωθεί και να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση. Ευχαριστώ η κυρία Χάουταλα για τους πρασίνους, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Ήπατη εκπρόσωπε, απηχείτε τα συναισθήματά μας απολύτως όταν λέτε ότι συγκλονιστήκατε. Συγκλονίστηκαν πράγματι μετά την 19η Δεκεμβρίου, διότι πολλοί από εμά ελπίσαμε ότι θα υπήρξε μια σταδιακή, ένα σταδιακό άνοιγμα της Λευκορωσίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα πολλές από τις ελπίδες για την ώρα έχουν εξαφανιστεί. Και είναι πολύ ανησυχητικό που ακούμε σχεδόν κάθε ώρα ειδήσει από το Μίνσκ και άλλα τμήματα της Ευκορωσίας για συνεχή μέτρα καταστολής χτες μάλιστα, είχαμε παρενόχληση κατά της Διέσνα, της Οργάνωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ε, συνεχίζονται επιδρομές κατοίκων, συλλήψεις, κρατήσεις και αυτή είναι μια οργάνωση η οποία ήταν ε, πολύ γενναία όσον αφορά την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία και δεν επιτρέπει να καταχωρηθεί, να καταγραφεί επισήμω το Μητρό από τι αρχέ. Και η Επιτροπή Ζήχη τη Λευκορωσία πήρε μια προειδοποίηση, αφού ήταν σε επαφή με τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την εξαρτησία των δικαστών και των νομικών, διότι πιστεύουν, έχουν λόγο να πιστεύουν ότι αυτοί που έχουν ε, κατηγορηθεί με πολύ ε, βαριές κατηγορίες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να δικαστούν δίκαια. Ε, επίσης, ακούμε σήμερα ειδήσει για την ε, πρώην υποψήφιο πρόεδρο κ. Σάνικοφ και τη σύζυγό του που δημοσιογράφο ανταποκριτή της Νοβάγια Γκαντζέτα την Ειρήνα Χάλεπ στο Μίνσκ και για το παιδί τους που προξάνε σε αίσθηση σε όλο τον κόσμο δηλαδή ίσως το παιδί μπορεί να μείνει με τους παππούδες όσο κρατούνται οι γονείς αλλά σας προειδοποιώ αυτή δεν είναι τελική καλή είδηση περιμένουμε επιβεβαίωση που ίσως να έρθει την επόμενη εβδομάδα γιατί ε, γιατί συμβαίνουν αυτά, αυτή η καταστολή, αυτή η καταπίεση στη Λευκορωσία. Πρέπει να επιμείνουμε επί της ανεξάρτητης διεθνούς έρευνας για τα όσα συνέβησαν, να καταλάβουμε ποιο είναι το ιστορικό, τους λόγους, να καταλάβαμε αν υπήρξαν κάποιοι που προκάλεσαν, ε, α, ξεκίνησαν αυτά τα βία γεγονότα. Και θεωρούνται κλιματίες αυτού που ζητούσαν δημοκρατία στην ε, Λευκορωσία τώρα. Και καταλήξαμε. Ο πιο ενδεδειγμένο φορέα για τη διεξαγωγή τέτοιων ερευνών θα ήταν ο ΑΣΕ και αν όχι αυτό ο φορέα, τότε τα Ηνωμένα Έθνη. Τι, τι θα λέγαμε για νέε εκλογέ, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν ζητούμε να διεξαχθούν γρήγορα νέε εκλογέ, διότι θα πρέπει να μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα εφαρμοστεί ο δικό χάρτη δημοκρατικέ μεταρρυθμίσει. Πρέπει να εγγυηθούμε την ελευθεροτυπία, ε, την ελευθερία ε, τη συνέλευση χωρί μέχρι ότου να μπορέσει να, διεξα... να διεξαγάγει η Λευκορωσία νέες εκλογές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να σκεφτούμε αν πρέπει να κατηγορήσουμε εκτός από τους ίδιους τους Λευκορώσους κυρίως να κατηγορήσουμε και τους εαυτούς μας. Και κοιτάξτε να δείτε τι άλλες περιπτώσεις όπως τον Πρελουσκόνη και άλλες. Και, και έτσι έρχεται να νομιμοποιηθεί το καθεστώς το λευκορωσικό. Σικόρσκι, Βέστερ Βέλε, οι ενέργειές τους νομιμοποιούν το καθεστώς του Λουκασέγκο. Οι πολιτικοί, οι πολιτικάντιδες κάθονται και δημιουργούν ευμενείς συνθήκες για να έχει περιθώριο λιγμόνο ο Λουκασέγκο, χωρίς να του ζητάνε τίποτα. Επομένως, κατηγορούμε τη Λευκοσία, αλλά να κατηγορούμε τους εαυτούς. Κύριος Σόλτς, για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, η δική μου κοινοβουλευτική ομάδα <clears throat> δεν έχει υπογράψει τη συμβαστική πρόταση ψηφίσματος για τη Λευκορωσία. Θέλω όμως ρητά να πω ότι αυτό δεν πρέπει να εμεινευθεί ότι το αποτέλεσμα των εκλογών τη σύλληψη και την δίωξη των αντιφρονούντων στη Λευκορωσία τη δεχόμαστε. Για μένα, για μας δίκαιες και ε, δημοκρατικές εκλογές καθώς επίσης και η ελευθερία των άλλων είναι σημαντική υπόθεση. Αναφέρω παράθεμα της ε, Ρόζα Λούξεμπουργκ. Αυτό είναι η θέση μας ε, και σε σχέση με τη Λευκορωσία και σε άλλες χώρες. Η άμεση απελευθέρωση όλων των κρατουμένων και φυλακισμένων. Αμφισβητώ όμω, αμφιβάλλω, αν κυρώσει είναι ένα σωστό μέτρο για να απελευθερωθούν άμεσα οι κρατούμενοι και η δημοκρατία στην Λευκορωσία να μπορέσει να επιβληθεί. Οι κυρώσει ήδη και στο παρελθόν είχαν επιβληθεί και στην Λευκορωσία Λευκορωσία και αλλού, αλλά δεν είχαν δώσει αποτελέσματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, το γνωρίζετε αυτό όπως και εγώ <clears throat> πολιτικά υπεύθυνα για σε ένα πολιτικό διάλογο με τα δικά μας αιτήματα πρέπει να αντιπαρατεθούμε με τους ε, Λευκορώσους με την επισήμανση για τις επικρίσεις και σε σχέση με την ε, ε, κοινωνία των πολιτών που προσπαθεί το καθεστώς να υπονομεύσει. Και έτσι σε σχέση με την ε, συνάφεια και συνεκτικότητα των δικών μας διαβημάτων η συνεκτικότητα αυτή είναι η καλύτερη οδός πιστεύω και η πιο έντιμη οδός ώστε τα δικά μας επιχειρήματα να εισακωστούν σε σχέση και με την σημερινή πρωινή συζήτηση για την Ουγγρική Προεδρία. Αυτό αποδεικνύεται. Ευχαριστώ. Για την Ευρώπη Ελευθερίας Δημοκρατίας για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αυτή η βίαιη καταστολή οποιασδήποτε εναλλακτική από τις 19 Δεκεμβρίου που έγιναν οι εκλογές είναι κάτι το οποίο έχει μειώσει το περιθώριο για τις ξένες δυνάμεις και αυτό έχει να κάνει και με τη σχέση Μίνσκ-Μόσχας τελευταία διετία τριετία. Γιατί ο Λουκασέγκο προς τα εκεί αληθορίζει από ό,τι χρειάζεται να μπει περισσότερο το ευρωπαϊκό στοιχείο, η ευρωπαϊκή πολιτική στην κοινωνία της ε, χώρας. Χρειάζεται να δείξουμε βέβαια πριν γίνει οτιδήποτε άλλο η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Χρειαζόμαστε επίσης να κάτσουμε και να συζητήσουμε για μια στρατηγική με την αντιπολίτευση στη χώρα. Αλλά πρέπει και να παρακολουθούμε στενά την συμπεριφορά της εξουσίας εκεί, αλλά μην αφήσουμε με τίποτα να πέσει η χώρα στα νύχια της Κίνας ή της Ρωσίας. Ε, ο κύριος Ογκουρεάνου για 1,5 λεπτό. Thank you, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Αλεξάνδρε Λουκασένκο ποτέ δεν έχασε την ευκαιρία για να αποδείξει ότι είναι δικτάτορ. Οι εκλογές του Δεκεμβρίου ήταν μια τελετή επαναδιορισμού. Αλλά εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουμε στην αυταπάτη ότι θα αλλάξει ως διαθαύματο ο Λουκασένκο. Και πράγματι είπαμε ας περιμένουμε για τι δεκεμβριανές εκλογές. Ε, ήρθαν οι εκλογές και ο Λουκασένκο παραμένει ίδιο και η αντιπολίτευση είτε είναι στο νοσοκομείο είτε στη φυλακή. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να επανεξετάσει την προσέγγιση τη όσον αφορά τη Λευκορωσία. Σαφώ δεν υπάρχει χώρο για τη Λευκορωσία στην εταιρική σχέση συνεργασία. Ε, θα πρέπει να ανασταλεί αυτή η σχέση. Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να είναι ο μόνο μα εταίρο. Περιμένω το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων τη 31η Δεκεμβρίου και η κυρία Ηλέδη Άστον και επίτροπος Φούλε, ελπίζουμε να προτείνουν αναστολή. Θα πρέπει να είμαστε ε, ειλικρινεί στην προσέγγιση μας. Δεν μπορούμε να δώσουμε βέτο για το Euronest όσον αφορά το Λουκασένικο. Χρησιμοποίησαν το Euronest για να μπλοκάρουν τη λειτουργία του. Το Euronest θα πρέπει να ξεκινήσει λοιπόν κατεπηγόντω μάλιστα. Ο κύριος Παλέκης για δυόμιση λεπτά. Σα ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ψηλή, εκπρόσωπε, θα πρέπει νομίζω να είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που θα στείλετε στην Δευκροσία, ε, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, όσο δεν είναι ακόμα αργά, θα πρέπει να επανέλθουμε και στο καθεστώ το οποίο ίσχυε πριν τι 19-12. Θα πρέπει να κινητοποιηθούμε, ούτω ώστε να ε, ακολουθήσουμε την, την, ατραπό ε, του, των δειγμάτων ανθρώπου, της λογικής, του δικαίου. Και σήμερα το πρώτο θέμα είναι το πώς να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι. Και θα πρέπει να υπάρχει η, η, η αίσθηση η οποία να σταματήσει αυτούς τις καταστολές κατά του τύπου κατά του, του, του πολιτικού κόσμου. Επομένω, βέβαια, δεν θα πρέπει να τιμωρήσουμε τον κόσμο. Να είμαστε προσθετικοί στα όσα θα κάνουμε και να αποφύγουμε το να τιμωρηθεί, να υποστεί τι κυρώσει ο κόσμο, γιατί ταυτόχρονα θα πλήξουμε και τι οικονομικέ, πολιτικέ, επιστημονικέ σχέσει μα με τη χώρα. Χρειάζεται όλα αυτά να τα διατηρήσουμε γιατί θα ανοίξει η κοινωνία η δε πολιτική του διαλόγου με την χώρα αυτή τα τελευταία χρόνια έτσι όπως έγινε νομίζω ότι έχει αποδώσει κάποιους καρπούς σήμερα δε έχουμε 50% των Λευκορώσων οι οποίοι είναι υπέρ στο να υπάρχουν πιο στενές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιδράσουμε μετά όσα έχουν γίνει στο Μίσκ με τέτοιο τρόπο ούτω ώστε οι φιλοευρωπαίοι όχι μόνο να μειωθούν αλλά και να αυξηθούν. Να μην είναι επώδυνες δηλαδή οι που επιβάλλουμε ως προς τους ε, οργανωτάς των εκδηλώσεων που και γίνονται και τώρα όσον αφορά το αυτό που λέμε το τείχος του Βερολίνου για θεωρήσεις και άλλα θέματα πρόκειται ότι για έναν τείχο ο υπάρχει μεταξύ Ευρώπης και των γειτόνων της προς Ανατολάς υπάρχει αυτό και προς την Λευκορωσία ήρθε η ώρα να γκρεμίσουμε και αυτό το τείχος ούτως ώστε να υπάρχουν εύκολα προσβάσιμες θεωρίες διαβατηρίων για όλους τους πολίτες της Ουκρανίας, της Γεωργίας, της Ρωσίας, της ε, Λευκορωσίας. Μιλάμε για ένα εκατομμύριο ευρώ τα οποία μαζεύουμε για από τις βίζες είναι πάρα πολλά λεφτά, υπερβολικά. Και πού πάνε όλα αυτά, δεν πάνε για να γεφυρώσουν το χάος μεταξύ της Ένωσης και των, γειτόνων της Ανατολής. για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε. και στην πολιτική και στη ζωή μετράει πάρα πολύ η ελπίδα, οι προοπτικές, οι προσδοκίες για μια βελτίωση στο μέλλον. Η ελπίδα είναι αυτό που 19-12 εξαφανίστηκε από τη χώρα. Α ελπίσουμε ότι οι επόμενε εκλογέ θα είναι πιο δημοκρατικέ και α ελπίσουμε ότι η αντιπολίτευση θα μπορέσει να κατέβει στι εκλογέ και ότι τα μέσα ενημέρωση θα μπορέσουν να αποτυπώσουν το πολιτικό σκηνικό προ τον κοσμάκι. Όλα αυτά τώρα δεν ισχύουν, άρα θα πρέπει να αλλάξουν την πολιτική μας προς τη χώρα. Χρειάζεται μια προσέγγιση θετική, είχαμε πει, χρειάζεται ένα άρα μια, θετική στάση και προσέγγιση. Δεν απέδωσαν όλα αυτά. Άρα θα πρέπει να δούμε τι κυρώσεις θα επιβάλλουμε, αλλά να δούμε πώς θα σταματήσει η διαπλοκή στη χώρα, Ίσως ε, προς τα εκεί πάμε καλά γιατί η Κομισιόν ορθώ ζήτησε την ε, απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων άρα το συντομότερο δυνατόν θα πρέπει να στείλουμε αποστολή προς τη χώρα και να επιμείνουμε να υπάρχουν μη κυβερνικές οργανώσεις, κοινωνία πολιτών, ε, οργανώσεις αντίστοιχες να υπάρχουν και να τα πούμε και στους Ρώσους δεν έχουν προβληθεί όσο πρέπει τα προγράμματά μας για τη χώρα. Γεωργία, Αρμενία, Ουρμπανία, ε, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, όλες αυτές είναι χώρες που είναι σημαντικές και είναι χώρες που βρίσκονται κοντά στην Ευρώπη και όλα αυτά αν τα κάνουμε θα δώσουμε ελπίδα στη χώρα. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπάτη εκπρόσωπη, η ελπίδα μας ότι με τις προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία η χώρα θα το προς την δημοκρατία απογοητεύτηκαν πικρά. Παρόλες τις αρνητικές, τα αρνητικά αυτά βιώματα και τις επιφυλάξεις έναντι της κυβέρνησης Λουκασένκο, είχε τίνει ε, βίκονους ε, και χείρα βοηθείας η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Λουκασέγκο. Ήταν αδιαμφισβήτητα σαφής, αυτή η διαδικασία και σε σχέση με τις τις εκλογές που θα γινόντουσαν με τρόπο δίκαιο και δημοκρατικό. Όμως ε, έχουν τόσο κλονιστεί, τα, ε, ε, οδήγησαν σε τέτοιο κλονισμό τα γεγονότα που αναγκάστηκε να δείξει το πραγματικό του πρόσωπο ο δικτάτορας. Δεν νομιμοποιείται η εξουσία του και η βία κατά της αντιπολίτευσης είναι ένα έγκλημα. Αυτό είναι μια μεγάλη οπισθοχώρηση, οπισθοδρόμηση για την Λευκορωσία. Επικρατεί φόβος, τρόμος και σε σχέση με τους νοθευτές των εκλογών δεν είχαν αναμειχθεί διπλωμάτες άλλων χωρών αλλά οι ίδιοι ήταν υπεύθυνοι και σε σχέση με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται όπως και στην εποχή του Στάλιν από την τοπική ΚΑΚΕΜΠΕ την μυστική υπηρεσία και ένα, ε, σε σχέση με αυτό το μετακομμουνιστικό ε, καθεστώς είναι πραγματικά παράδεκτο και αφόρητο. Έχουμε προετοιμάσει ένα ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που αποτελεί καλή βάση για τη διαβούλευση των Υπουργών Εξωτερικών. Πρόκειται ω αιτήματα για την άμεση απελευθέρωση των κρατουμένων, την περίθαλψη των ε, τραυματισμένων και την άμεση λειτουργία μιας ε, ανεξάρτητης ε, επιτροπής διακρύβωσης των γεγονότων ώστε να δούμε τι θα μπορέσει να γίνει σε σχέση με αυτή την κατάσταση. Τώρα θα πρέπει να βοηθήσουμε τις φιλευρωπαϊκές δυνάμεις που δημιούργησαν, απέκτησαν ελπίδες ότι κάτι θα άλλαζε και που βλέπουν το μέλλον της χώρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι σε μια στενότερη δέσμευση προς τη Ρωσία. Και όταν βλέπουμε εδώ ότι ο Πρωθυπουργός, ε, ο Πρόεδρος Πούτιν, ε, ο ή ε, ο Λουκασένκο δείχνουν πώς κατανοούν την δημοκρατία και πιέζουν τη Λευκορωσία προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ξεκινήσω με πληροφορίες ε, για την κυρία Χαουτάλα. Ελπίζω ότι έχει τα ακουστικά της και μπορεί να παρακολουθήσει αυτά που θα πω. Οι πληροφορίες ε, για την οργάνωση Βέσνα θα πρέπει να συμπληρωθούν και από κάποια άλλη πληροφορία. Όχι μόνο δεν μπορούν να καταχωρηθούν σε Μητρώα, αλλά η αστυνομία δίμευσε, κατέσχε όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές τους και την Δευτέρα ήδη και όλα υπήρχε ε, συλλογή ηλεκτρονικών υπολογιστών για να αποσταλούν σε αυτή την οργάνωση. Σε σχέση τώρα με την Επιτροπή, πράγματι είναι χρόνος ε, να δράσουμε τώρα. Και ένα άλλο πράγμα, δεν πρέπει να απομονωθεί, δεν πρέπει να απομονωθούν οι Λευκορώσοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Ήπια μέτρα είναι αυτά τα οποία χρειάζονται. Η δημιουργία, η ανοικοδόμηση της κοινωνίας των πολιτών, για παράδειγμα. Η άρση των περιορισμών όσον αφορά θεωρήσεις διαβατηρίων για τους πολίτες αυτής της χώρας. Θα πρέπει αυτό παράλληλα να εξεταστεί με κάποια σκληρά μέτρα όπως προτείνονται από την κυρία Όιλαντ ή τον κύριο Ποτασέβιτς. Θα πρέπει να συνδυάζονται και η ήπια και η σκληρή αυτή προσέγγιση σε μία ενιαία προσέγγιση. Thank you. Ευχαριστώ. Είπατε εκπρόσωποι, νομίζω ότι η διάγνωση ε, που έχει γίνει και η θεραπεία που έχει προταθεί είναι ορθή και έχει προγραμματιστεί. Δεν είχαμε διαφορετική προσέγγιση στο παρελθόν, αλλά κάναμε ελάχιστα. Άρα πρέπει να διαρωτηθούμε. Είμαστε αρκετά αποφασισμένοι να κάνουμε κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Πρέπει να καταδικώσουμε και να ζητήσουμε απελευθέρωση, να επιβάλλουμε κυρώσεις, να εξετάσουμε το δεχόμενο στολής διακοπής των συμφωνιών. Εάν δεν προχωρήσουμε από την ηθική υποστήριξη και τα ρητορικά σχήματα, δεν θα έχουμε καρπούς. Χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμη δράση και αυτή θα είναι η δοκιμή για την νέα εξωτερική πολιτική που θέλετε να ακολουθήσετε, λέει διάστον. Και δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τη Λευκορωσία. Πώ θα αντιμετωπίσουμε το θέμα τη Λευκορωσία θα αποφασίσει την γεωπολιτική δυναμική περιοχή. Μολδαβία, Ουκρανία, Ρωσία και Αλαχού. Για την ώρα η Λευκορωσία απομακρύνεται από την Ευρώπη και αποσύρεται και από την Ουκρανία η Ευρώπη. Χρειάζεται διτή προσέγγιση, κυρώσεις, άνοιγμα της κοινωνίας. Χρειάζεται να αυξήσουμε τη βοήθεια κλπ. Να αντικαταστήσουμε την πολιτική διαφόρων κινήτρων και ποινών που κοθήσαμε μέχρι τώρα ε, όσον αφορά το καθεστώ, αλλά να κάνουμε κάτι τέτοιο ανά της κοινωνίας. Αλλά εταίρος μας είναι η κοινωνία και όχι το καθεστώς. Αυτό πρέπει να θυμόμαστε. Κυρία Άστον, είπατε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθούμε. Θα πρέπει να, κάνουμε τόσο να συνεχίσουμε να κάνουμε τόσα λίγα όσο κατά το παρελθόν. Κάναμε όλοι όσα θα έπρεπε να κάνουμε, όχι. Ήτανε... Η βοήθεια ήταν γελιοδός μικρή. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάουιτ ε, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε συζητούμε σήμερα και φαίνεται ότι ο Λουκασέγκο τελικά ε, θα, θα αναλάβει τα καθήκοντά του την Παρασκευή χωρίς να υπάρχουν ε, φιλοξενούμενοι ξένοι. Θα αναλάβει τα καθήκοντά του. Η εθνή κοινότητα δεν αναγνωρίζει τι εκλογέ τη Λευκορωσία ότι ήταν δίκαιε, ελεύθερε και διαφανεί. Εάν το κάνει αυτό, θα είναι μια μαύρη Παρασκευή να ακολουθήσει την αιματηρή Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου, όταν 700 δημοκρατικοί διαδηλωτέ ε, και νέοι υποψήφοι ε, ε, δέχτηκαν, ξυλοδάρθηκαν, αλλονού του πάσαν τα πόδια, Κάποιο έπαθε κεφαλικά, βλάβε βλάβες και ζητώ από τα κάτι μέσα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και την είπατε εκπρόσωπο να υποστηρίξουν την πολωνική πρόταση για απαγόρευση θεωρήσεων και όπω λέει το ψήφισμα να προστομίσουμε την αρχή για περαιτέρω εστιασμένε οικονομικέ ποινέ. Και ένα από τα πράγματα που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να εκφράσει σαφή αιτήματα, απλά αιτήματα για την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, οι αρχές να άρουν απειλή περιορισμού της Επιτροπής Ελσίνσκη, Επιτροπής Ελσίνκη της ε, και να διοργανωθούν γρήγορα ελεύθερες εκλογές. Για το μέλλον συμφωνώ με τα υποθέντα, αυτά που είπε κάθε Άστον και η ομάδα μου. Πρέπει η πολυμερής προσέγγιση παραμείνει ανοιχτή και να τονίσουμε την προσέγγιση κοινωνία των πολιτών και να την υποστηρίξουμε. Δεν είναι θέμα μόνο δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Λευκορωσία. Είναι και μια δοκιμασία για την πολιτική γειτονία τη Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Χρειάζεται στενότερη συνεργασία με τους γείτονε για να θαρρύνουμε διαδικασία προσέγγιση στη δημοκρατία και προσέγγισης μεταξύ μας. Δεν θα λειτουργήσει αυτό αν λείπουν αμοιβέ δεσμεύσει, έλλειψη δρά... όταν δεν σέβονται τι υποχρεώσει και γίνονται... υπάρχουν προβλήματα. Δεν θέλουμε απλώς ευφυείς ποινές κατά της Λευκορωσίας. Θέλουμε να αποφύγουμε το φυσικό πόνο που δέχονται οι άνθρωποι που δέρνονται. Εμείς υποστηρίζουμε τη δημοκρατία και τα ανθρωπίνα δικαιώματα όπως και αυτοί. Πρέπει να σταθούμε στο πλευρό τους, σε αλληλεγγύη. Ούτω ώστε επιτέλου να περάσουν τα μακρά χρόνια τη βασανιστήριων για τη Λευκορωσία. για λεπτά. Αξιότιμη είπατε εκπρόσωπο. Σας ευχαριστώ για την ταχεία αντίδραση στα γεγονότα στο Μίνσκ. Επίσης σας δίνω και την αναγνώρισή μου για την προσέγγιση σας ότι πρέπει ισόρροπα να δράσουμε σε σχέση με τις κυρώσεις έναντι των υπεύθυνων για τις ε, σοβαρές αυτές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε σχέση με μέτρα που θα ληφθούν υπέρ των πολιτών της Λευκορωσίας. Θα ήθελα από αυτή τη θέση να εκφράσω ευχαριστίες ε, για την διάσκεψη για την ασφάλεια στο Μόναχο που ε, είπαν ότι δεν ήθελαν τον Λουκασέγκο ανάμεσά τους και δεν τον προσκάλεσαν. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι οι δικτάτορες δεν είναι πρόσδεκτοι σε διεθνή φόρα διότι η διεθνής ε, ε, αναγνώριση ενός αυτόκλητου Προέδρου <clears throat> δημιουργεί μια, ας το πω έτσι, εντός εισαγωγικών διεθνή αναγνώριση των μη δημοκρατικών εκλογών. Γι' αυτό αυτή η αντίδραση ήταν η απόλυτα σωστή αντίδραση, να μην προσκληθεί ο Λουκασέγκο εκεί. Για πολιτικές αλλαγές στην Λευκορωσία πρέπει μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ένα μεγάλο χρονικό ορίζοντα να έχουμε με μακροπρόθεσμες προοπτικές όμως για την ανθρωπιστική κατάσταση στην ίδια τη Λευκορωσία, κυρία Άστον, δεν πρέπει να αναμείνουμε περισσότερο και να σταυρώσουμε τα χέρια μας. Πρέπει αμέσως να αντιδράσουμε και να διασφαλίσουμε άμεσα ότι θα απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι. Οι θα μπορέσουν τα παιδιά να επιστρέψουν στους γονείς τους και τα παιδιά να ξαναβρούν τους γονείς τους γιατί δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να αγωνιστούν και να διαδηλώσουν για τα δημοκρατικά δικαιώματα και να καταστήσουν σαφές με τις διαδηλώσεις στους δρόμους ότι αυτά ήταν τα αιτήματά τους. Η αντίδραση απέναντί τους ήταν πραγματικά υπερβολική και αθέμητη και θέλω να διασφαλίσετε με κάθε κάθετο τρόπο ότι πρόκειται για πολιτικούς κρατούμενους και όχι για εγκληματίες. Και χαιρετίζω τον Αντρέ Σάνικοφ και τους άλλους όλους που βρίσκονται ω κρατούμενοι ε, στι φυλακέ, είναι φυλακισμένοι. Πρέπει να ξέρουν ότι έχουν την αλληλεγγύη μα στο πλευρό του. Του υποστηρίζουμε. Υψηλή εκπρόσωπε, επίτροπε, συνάδελφοι, πριν από ένα χρόνο δεν άφησαν τον Φαρίνας να έρθει εδώ στο Στρασβούργο να παραλάβει το βραβείο Ζαχάροφ. Αυτό έγινε από ένα ε, καθεστώ προσβλητικό όπω το σημερινό του Λουκασέγκο που σήμερα ε, είναι τόσο αυταρχικό. Είναι αυταρχικό, ήταν ολοκληρωτικό τη Κούβα, αλλά τέλο πάντων σήμερα θα πρέπει να δούμε πώ θα σταματήσουμε την Λευκορωσία με τέτοιο καθεστώ να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποτέ δεν είχε η χώρα ελευθερία και δημοκρατία. Βέβαια οι πολίτες της χώρας είναι ευπρόσδεκτοι. Όμως οι εκπρόσωποι του καθεστώτος Λουκασέγκο θα πρέπει να τους αφήσουμε απ' έξω. Και αυτό γιατί δεν δίνουν κανένα σεβασμό προς την κοινωνία και το, τη δημοκρατία. Κούρσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόσφατα κάποιες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ακολουθούν κάποια συγκεκριμένη πολιτική προ την Λευκορωσία. Το ίδιο ισχύει και για την κυβέρνησή μου. Πρώτοι για πολιτικέ που απέφυγαν. Ο Λουκασέγκο, που είναι ο τελευταίο Ευρωπαίο δικτάτορα, φυλακίζει του πολιτικού του αντιπάλου. Η πολιτική τη συμφιλίωση δεν έχει αποδώσει αποτελέσματα. Επομένω, αυτέ μα οι κινήσει εξελίχθησαν ω υποστήριξη προ τον Λουκασέγκο, ο οποίο συνέχισε την άσκηση βία κατά των πολιτικών αντιπάλων. Η Ευρώπη πρέπει να δείξουμε ότι δεν θα ανοιχθεί περαιτέρω καταστολή των πολιτικών ελευθεριών. Να τιμωρήσουμε βέβαια το καθεστώς και όχι τους πολίτες της χώρας οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια και η αντιπολίτευση και τα μέσα ενημέρωσης επομένως θα πρέπει ή να σταματήσουμε ή να αναβαθμίσουμε την συνεργασία μας, την εταιρική με τη χώρα δεν θα πρέπει αυτό το καθεστώς να δει ούτε μια δεκάρα από μα για να καταρρεύσει. Αδελφοί, τώρα περνάμε στην διαδικασία του Catch the Eye. Πρώτα ο κύριο Κέλλη, θα είμαι αυστηρό στην ώρα, είναι πολλοί ομιλητέ, για ένα λεπτό. Ε, Νομίζω ότι μία από τις μεγάλες εξελίξεις στο σύγχρονο κόσμο είναι η μετάβαση από ολοκληρωτισμό στη δημοκρατία στην Ανατολική Ευρώπη, στις χώρες Ανατολικής Ευρώπης. Ουγγαρία με τον πρόεδρο της οποίας, με τον υπουργό της οποίας συζητήσαμε το πρωί ήταν ένα παράδειγμα και ο πρόεδρός μας ο κ. Ζιμπούζεκ είναι ένα λαμπρό παράδειγμα αυτών των εξελίξεων όμως υπάρχουν και άλλες χώρες όπου η μετάβαση δεν ήταν ομαλή η Λευκορωσία δυστυχώς είναι τέτοιο παράδειγμα και ιδιαίτερα η Λέδη Άστον συνόψισε το τι θα πρέπει να γίνει όσον αφορά την αντιμετώπιση καταστάσεως. Το καλύτερο που μπορεί να πει κανεί είναι ότι έχουν αστερνιστεί την δημοκρατία μέσω δύο βημάτων προόδου και ενό ε, βήματο υπαναχωρήσεω. Στι πρόσφατε εκλογέ κάναν τρία βήματα προ τα πίσω και κανένα βήμα προ τα μπρο. Νομίζω ότι σωστά μα επιλεδιάστον ότι πρέπει να συνεργαστούμε με την κοινωνία των πολιτών, τι μη κυβερνητικέ οργανώσει και του διεθνού εταίρου μα, ούτω ώστε να ασκήσουμε πίεση στο Λουκασέγκο, ώστε να σταματήσει την καταστολή και την δικτατορία του. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Γκριζίμ, για ένα λεπτό. Σε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν η περιστολή, καταστολή της ίδιας της δημοκρατίας και των πολιτικών δικαιωμάτων και η σύλληψη τόσων πολλών πολιτών και των υποψηφίων για την Προεδρία που δεν χρειάζεται πραγματικά κανένα σχόλιο. Είναι μια δοκιμασία πραγματική αυτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τους εταίρους μας, για τους εταίρους που έχουν προ, ξεχωριστή ειδική σχέση μαζί μας, εταιρική σχέση όπως τη Ρωσία. Πρέπει να υποστηρίξουμε ε, το αίτημα ότι πρέπει άμεσα να απελευθερωθούν οι κρατούμενοι. Προτού ξεκινήσουν συνομιλίες με τους ε, ε κρατούντες στη Λευκορωσία. Θα πρέπει όμως ε, να λάβουμε υπόψη τους πολίτες και να αλλάξουμε το καθεστώς θεωρήσεων διαβατηρίων. Επίσης πρέπει να υποστηρίξουμε τους ε, φοιτητέ της Λευκορωσίας που θα πρέπει να γίνουν δεκτοί σε άλλα πανεπιστήμια, σε άλλες χώρες ε, και να υποστηρίξουμε επίσης την ελευθερία του τύπου την ελευθερία των τηλεοπτικών σταθμών και της τηλεόρασης και να εργαστούμε για αυτούς τους στόχους. Κύριε Πρόεδρε, είναι φανερό ότι στη λευκορωσία τα πράγματα έχουν εξελιχθεί πολύ άσχημα για τις, δικές μας αρχές και τα δικά μας πιστεύω. Ο Λουκασέγκο είναι στην ηγεσία της χώρας και η αντιπολίτευση βρίσκεται στη φυλακή. Άρα αναμένει κανείς από εμά να κινηθούμε στην κοινωνία των πολιτών που ορθά αναπτύχθηκε προηγούμενα ότι στην κοινωνία αυτή χαίρει εκτίμηση η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αρχές της να αναζητήσουμε την ελευθερία του τύπου την απελευθέρωση των φυλακισμένων αρχηγών της αντιπολίτευσης και πολύ περισσότερο να οικοδομήσουμε μια τέτοια πολιτική αυτή που αναφέρθηκε από την κυρία ashton η οποία με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε νέες συνθήκες για να, ξαναπλησιάσουμε τη λευκορωσία. ευχαριστώ. Ο κύριος οι προεδρικές εκλογές στην χώρα ήταν μια μεγάλη απογοήτευση για εμάς που παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα και είδα τον πρέσβη στο Λονδίνο με διαβεβαίωση ότι αυτή τη φορά όλα θα είναι διαφορετικά σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ. Όμως το, το, το, το ένστικτο, το ρεφλέξ του σοβιετικού ανθρώπου τελικά είναι το αυτό που επιβιώνει περισσότερο απ' όλα και τελικά όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούν παρά να γίνουν ουρές. Παρακαλώ να ξαναγίνουν, είπαμε, οι εκλογές με παρατηρητές ένωσης και επίσης η διεθνής κοινότητα να δώσει το πράσινο φως σε σχέση με τον εύρυθμο τρόπο διεξήγησης των εκλογών. Αλλιώς θα πρέπει να πάμε σε πάγωμα περισσότερο του Λουκασέγκο στο εξωτερικό αυτού των ε, εξωματούχων του και να ξεκινήσουμε κάποιες αυστηρές κυρώσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκ μέρους μου θα ήθελα να υποστηρίξω αυτά που είπε η κυρία Άστον για ισορροπημένη στάση έναντι της Λευκορωσίας και των όσων συμβαίνουν εκεί. Πολύ συχνά μιλάμε με συναισθηματισμό. Υπάρχει συναισθηματική φόρτιση και κάνουμε προτάσεις και εκφράζουμε ιδέες με το συναισθηματισμό. Μιλάμε για πολιτικούς κρατούμενους και φυλακισμένους, αλλά δεν έχουμε... Δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα των διαφόρων δικαστικών υποθέσεων που δεν έχουν ε, οδηγήσει σε κάποια ποινή, σε κάποια απόφαση. Άρα θα πρέπει να ακολουθήσουμε ισορροπημένη προσέγγιση. Εδώ και δύο χρόνια κάτι παρόμοιο είχαμε και στην ε, Λετωνία. Σε μία, λοιπόν, συνεδρίαση κανείς δεν αρνήθηκε ότι υπάρχει το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε. Όταν όμως ήρθαν οι διαδηλωτές και πετέθησαν κάτω του Κοινοβουλίου, ε, αντέδρασε η αστυνομία σε αυτήν την περίπτωση. Άρα, από πού προέρχονται τελικά τα χρήματα που πάνε στην αντιπολίτευση της Λευκορωσίας. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Κύριε για ένα λεπτό. Πρόεδρε, Λοιπόν, για τα μέσα του τύπου και πάλι η εισαγωγή των κυρώσεων όσον αφορά τον πρόεδρο Λουκασέγκο που είχαν χαλαρώσει πριν από δύο χρόνια θα ήταν λέει η παναχώρηση ότι οι τις προσπάθειες για προσέγγιση έχουν αποτύχει. Εγώ πιστεύω ότι πιο πριν είχαν αποτύχει αυτές οι προσπάθειες ε, το αργότερο κατά τις προεδρικές εκλογές ή με το κλείσιμο του γραφείου του ΟΣΑ, του ΑΣΕ στην ε, ε, Λευκορωσία. Η περίπτωση αυτή του τελευταίου δικτάτορα στην Ευρώπη δείχνει ότι έχει πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Ένωση με την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το σκάνδαλο με τη CIA, με τις ε, μυστικές ε, κρυφές πτήσεις ε, και όσον αφορά την, τα, θέματα της αυτοδιάθεσης κρατών, για παράδειγμα στη, στα Βαλκάνια την εικόνα του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχει αμαυρώσει. Η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπονομεύεται όταν βλέπουμε σε σχέση με την Τουρκία όταν συνεχίζονται διαπραγματεύσεις με μια χώρα δηλαδή που έχει τεράστια ε, κενά που πρέπει να καλύψει όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή την κατάσταση σε σχέση με τον Λουκασέγκο. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Καρινόφσκι για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, το καθεστώς Λουκασέγκο κλιμακώνει την καταστολή και άρα είναι καθήκον μας να δώσουμε ελληνική προς το λαό της χώρας. Να στηρίξουμε τα μέσα. Καλό παράδειγμα αυτό το οποίο είναι με την Πολωνία. Επίσης ε, υποτροφίες προς φοιτητές, αυτούς που διώχνουν τα πανεπιστήμια γιατί αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση είναι και αυτό ένα καλό παράδειγμα. Επίσης ε, θα πρέπει να φτηνίνει και η βίζα από τη Λευκορωσία και αυτό να αλλάξει και να τους επιτρέψουμε ελεύθερα να ταξιδεύουν ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως να εξαιρούνται οι εκπρόσωποι της κυβερνήσεως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν να βγαίνουν και να κυκλοφορούν οι εκπρόσωποι της κοινωνίας της Λευκορωσίας. Και έτσι θα γίνουν αλλαγέ στην κοινωνία και έτσι θα γίνει καλύτερη χώρα. Η κυρία Μπασέσκου για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Οι προεδρικές εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου είναι για μας ένα πισωγύρισμα και για την δημοκρατική εξέλιξη της χώρας αλλά και όσον αφορά τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βία αντιμετωπίζεται από την αντιπολίτευση ως πολιτικό όπλο και δεν, δεν υπάρχει δικαίωμα στην αντιπολίτευση να εκπροσωπηθεί στο κοινοβούλιο. Πρόκειται για ένα αυταρχικό καθεστώς το οποίο δεν θα έπρεπε να απολάβει των προνομίων της εταιρική σχέσης με τη Δύση. Ούτε έχουν δεσμευτεί όσον αφορά τις υποχρεώσεις του σε αυτή την εταιρική πολιτική όπως έκανε η Γεωργία και η Μολδαβία. Θα πρέπει να μπει ένα φρένο, θα πρέπει να μπει στο ψυγείο η χώρα αυτή όσον αφορά την εταιρική σχέση με την Ανατολή. Θα είναι αυτό ένα μάθημα προς την κυβέρνηση. Ελπίζω το επόμενο ε, Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής θα αποφασίσει εν λόγω. Σε ευχαριστώ πρόεδρε. Είπατε εκπρόσωπε, έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση που να απευθύνω προ την ε, Λέδη Άστον. Εσεί γνωρίζετε τι ε, έγινε στο Μπούζεκ όσον αφορά το Λεβαντόσκι και λοιπά το βράδυ της 19ης Δεκεμβρίου έβαζαν το ραδιοσταθμό στο Radio Free Europe, στο BBC ή σε άλλους σταθμούς ε, για να μάθουν από αυτούς τι γινόταν. Και ένα άλλο θέμα, πώς κατάφερε ο Λεκ Βαλένσα να επιβιώσει, πώς μπορούσαν οι ηγέτες της αντιπολίτευσης που ήταν ε, ε, που εδιώχθησαν μπόρεσαν να επιβιώσουν κατάφεραν να επιβιώσουν επειδή οι συνδικαλιστές από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες τους βοήθησαν και τους υποστήριξαν και άκουγαν αυτούς τους ραδιοσταθμούς ε, επειδή υπήρχε χρηματοδοτική υποστήριξη για αυτούς τους σταθμούς. Τώρα είναι δική μας ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι οι Λευκορώσοι θα μπορούν να ακούσουν την αλήθεια και θα τύχουν και χρηματοδοτικής υποστήριξης για να μπορέσουν να ακούσουν αυτή την αλήθεια. Λέει Άστον, κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ απόλυτα με του συναδέλφου και προτείνω καλό καθεστώ του κασέν που κυρώσει και να δώσουμε υποστήριξη στην αντιπολίτευση τη Λευκορωσία, μη κυβερνητικέ οργανώσει και του απλού πολίτε. Το κοινό, η κοινή πρόταση ψηφίσματο αναφέρει ενδεχόμενη μετακίνηση του 2014 του Παγκοσμίου Κυπέλου στο ΣΥΝΚΙΑ από τη Λευκορωσία, αν δεν απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι λογικό εργαλείο, αποτελεσματικότατο εργαλείο. Αν ο Λουκασέγκο, ε, για το χόκι το πρωτάθλημα. Και το ίδιο είναι και οι πολίτε Λευκορωσία. Και αν μεταφερθεί το πρωτάθλημα του χόκι, θα δημιουργηθούν πολλά ερωτηματικά στη χώρα. Λοιπόν, ε, ε, ο αρμόδιο φορέα πρέπει να πάρει αυτή την απόφαση. Άρα θα μπορούμε έτσι να, να βελτιωθεί η εικόνα του. Διότι δέχτηκαν ε, πρώην αξιωματούχο του Κάτζομπέ και κομμουνιστή κατάσκοπο της ΚΑΤΖΕΜΠΕ στην ε, Αμερική και που έχει αρπάξει δισεκατομμύρια δολάρια. Η IHF ελπίζουμε τελικά να πάρει ε, τη σωστή απόφαση όσον αφορά αυτό το πρωτάθλημα. Η κυρία ε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι καλό που συχνά έχουμε εγκρίνει εδώ την αέκληση προ τη Λευκορωσία να γίνουν αλλαγέ. Δυστυχώ δεν λειτουργήσαν όμω αυτέ οι εκκλησει, δεν έδωσαν αποτελέσματα και έχουμε ένα πρόγραμμα εταιρική σχέσεως με αυτή τη χώρα που εμπεριείχε διάφορα ωφέλη οικονομικά και πολιτικά για τη Λευκορωσία και ήταν επιτυχής η πολιτική μέχρι κάποιο βαθμό, αλλά όπω είπε και ο κύριο ε, Ρούμπικ, αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι βοήθεια από το εξωτερικό για την αντιπολίτευση στην ε, Λευκορωσία. Αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι να εφαρμόσουμε κυρώσεις κατά της πολιτικής ηγεσία της Λευκορωσίας, αλλά να μην πλήξουμε τους πολίτες της χώρας που δυστυχώς έχασαν τόσα πολλά κατά τη διάρκεια των δημοκρατικών εξελίξεων. Χάσαν τη δυνατότητα να σπουδάσουν στο εξωτερικό, να εργαστούν στο εξωτερικό. Πρέπει να σταθούμε στο πλευρό του λαού της Λευκορωσίας και της μάχης που δίδουν για να πετύχουν τη δημοκρατία και την απαλλαγή στην δικτατορία. Ευχαριστώ. Okay, finally. Uh, Συνάδελφοι, να σας πω ότι θα το εκτιμούσα. Εκείνοι που ζητάτε να, να προσελκύσετε την προσοχή του Πρόεδρου, να είστε παρόντες στο θέατρο να μιλήσετε. Ο κύριος Μπόρις, για ένα λεπτό. σε ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι η ώρα της αλήθειας και της έκφρασης αλληλεγγύης προς τη Λευκορωσία. Είναι η τελευταία δικτατορία στην Ευρώπη αυτή η χώρα και γι' αυτό πρέπει να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς τους πολίτες της Λευκορωσίας. Και παρότι τα κονδύλια είναι ε, περιορισμένα σε σχέση με την υποστήριξη θα πρέπει να αναλυθεί ένα σοβαρό πρόγραμμα υποστήριξης για την αντιπολίτευση και τα μέσα ενημέρωσης και τους νέους εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές και πολίτες που δεν μπορούν να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια από πλευρά των Λευκορώσων. Θα έπρεπε να προετοιμαστεί ένα ειδικό πρόγραμμα έρασμος που θα ε, στοχοποιεί ιδιαίτερα τους ε, φοιτητές της Λευκορωσίας και θα είναι τέτοιας, τέτοιου είδους αυτό το πρόγραμμα που θα μπορεί με περιορισμένα κονδύλια να λειτουργήσει και θα είναι πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα που θα έχει για τον εκδημοκρατισμό της χώρας. η κυρία ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστώ και όλους τους αξιωτήμους βουλευτάς οι οποίοι έλαβαν μέρος σε αυτήν την τόσο σημαντική, εστιασμένη, ε, εις βάθος σημερινή συζήτηση και νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη πρόκληση το θέμα που θίγει το ψήφισμά Πέρασε πάνω από ένας μήνας, ε, όμως τα γεγονότα εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα και νομίζω ότι ήδη είμαστε σε θετική κατεύθυνση ακριβώς όπως όλοι επιθυμούμε να απελευθερωθούν οι κρατούμενοι και να είναι δυνατόν ε, όλοι οι φορείς της κοινωνίας εκεί να προχωρήσουν προς μια μεταρρύθμιση να συνεχιστεί η συνεργασία θέλουμε να μπορούμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο στο προτσές αυτό και όπως είπαν πάρα πολλοί βουλευτές αυτό το οποίο τονίσαμε στην αρχή είναι ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το πόσο είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο συνέβη θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι πρέπει να αναλυφθούν ε, ενέργειες προς εκείνη την κατεύθυνση, όμως ταυτοχρόνως πρέπει να βοηθήσουμε φοιτητές, μήντε κοινωνία των πολιτών, ε, όλους αυτούς για τους οποίους μιλήσατε κι εσείς και αν μου επιτρέπετε θα θεωρήσω ότι αποτελεί μεγάλη βοήθεια η στήριξη μέσω των όσων είπατε και κατακλείδη όταν πήγα και σαν τις οικογένειες των κρατουμένων αντιπολιτευτών ε, μου είπανε ότι είναι ξεκάθαρες οι προσδοκίες τους. Ε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε τόσο να απελευθερωθούν και να μπορέσει η χώρα να κάνει προ τα εμπρό, προ μια αυθεντική δημοκρατία όπω ανέκαθεν θέλαμε και αυτά τα είπα ε, προ τον Υπουργό Εξωτερικών. Ξεκάθαρα πάντω ε, είναι στα, στο χέρι τους να κάνουν αυτό. Πρέπει να αναστρέψουν το ρεύμα, οπότε θα πρέπει και βέβαια και οι διεθνή κοινότητα να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έλαβα έξι προτάσει ψηφίσματο ε, για την περάτωση αυτή τη συζήτηση. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαρθεί αύριο στι 12 το μεσημέρι. Κυρία είπατε εκπρόσωπε, από τις 3 ώρες σε αυτή την αίθουσα. Τώρα είναι 6 και 4. Θέλετε να κάνουμε διάλειμμα 5 λεπτό για να χαλαρώσετε, από εσάς εξαρτάται, μπορούμε να συνεχίσουμε αν θέλετε. Πέντε λεπτά. Όχι, θέλετε να συνεχίσουμε. Ωραία, καλώς. Το είχατε προβλέψει το πρόβλημα αυτό. Yes, absolutely. Κύριε Αντιπρόεδρε, να πω ότι πρέπει να ταξιδέψω, να πάω στην Τουρκία για συνομιλίες για το θέμα του Ιράν. Ο Στέφαν Φούλερο, συνάδελφος και φίλος, θα συμμετάσχει στο επόμενο τμήμα της Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της κυρίας Γκόμες, Συμφωνία Πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιβύης.